Ladies and gentlemen, please take your seats. Καθίστε παρακαλώ. The next point of our agenda. Το επόμενο σημείο είναι η εξέταση της έκθεσης για τον ε, αντίκτυπο ε, των εξελίξεων σε ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές επί των ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας ε, στην Ευρώπη. Η Άννα Γκόμες είναι η συγγήτρια. Θα αρχίσουμε αμέσως με την εξέταση έκθεση. Κυρία Γκόμες, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα εξ αρχής να τονίσω πως ε, το αντικείμενο της έκθεσης είναι ο αντίκτυπος των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές ε, επί των ικανοτήτων ασφάλεια και άμυνα σε σχέση με το πακέτο που ονομάζεται το 2009. Δεν πρόκειται για τον αντίκτυπο στην ενιαία αγορά, του θα το αφήνουμε στους συναδέλφους στη ΣΥΜΚΟ. Το κείμενο των συναδέλφων σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση ε, με αυτή που επέλεξα και εγώ για την ε, έκθεσή μου. Το εφαλτήριο είναι μια αξιολόγηση των οδηγιών για το αμυντικό πακέτο ε, το 2009. Πιο συγκεκριμένη εφαρμογή τους είναι αποδυναμωμένες, δεν υπάρχει ενθουσιασμός, δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή και είναι πολύ αργή η διαδικασία. Θα συντάξει μια έκθεση του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή αυτών των ειδικιών και ελπίζω με τις εκθέσεις μας να συμβάλλουμε κι εμείς στη συζήτηση όπως εξάλλου και θα τροφοδοτήσουμε, το ελπίζω, ε, τις συζητήσεις που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα. Άπειρες φορές ε, έχει τονίσει το Κοινοβούλιο ότι οι μη συντονισμένες και ε, βαθύτατες περικοπές ε, στον προϋπολογισμό επηρεάζουν αρνητικά την αμυντική βιομηχανία και αποθαρρύνουν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής τεχνολογικής βάσης ε, εμποδίζοντας έτσι και την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας αλλά και την ασφάλεια εφοδιασμού ως προς τον εξοπλισμό στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη στρατηγική αυτονομία σε σχέση με τα προηγούμενα δέκα χρόνια λόγω των ε, κινδύνων, των προκλήσεων ε, στις οποίες ε, καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε. Έχει, έχει πιάσει φωτιά η, έχουν πιάσει φωτιά οι γειτονικέ μας χώρες, έχουμε απειλές όπως η τρομοκρατία, πολλές σειράξεις ε, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δώσει απαντήσεις ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. και να εξασφαλίσει, να, να, να, θωρα, ε, να, να θωρακιστεί η ο κύριος Τάραντ είπε ε, νωρίτερα ότι χρειαζόμαστε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Πέραν αυτού, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να υπερβούμε τις ε, δυνατότητες που μας δίνουν οι συνθήκες ε, και να υπερβούμε αυτές τις ενισχύει οδηγίες το 2009 και η ρίστον παρόδο τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν αυτές τις οδηγίες και όταν τις εφαρμόζουν ε, ε, είναι υπερβολικά αργή η διαδικασία και δεν ε, υπάρχει συμμόρφωση, απόλυτη συμμόρφωση με τις διατάξεις. Να υπερβούμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο ούτως ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών, να τους προστατεύσουμε, να φροντίσουμε για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, μιλούμε για στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται και συνδυασμός ε, του πολιτικού και στρατιωτικού δυναμικού. Ε, και αυτό είναι το ωραίο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Βλέπουμε ότι μετά την οικονομική κρίση, αντί να επιτυγχάνουμε το στόχο των οδηγιών του πακέτου ε, του 2007, δηλαδή να ενισχύσουμε το δυναμικό μας ε, και τη στρατηγική μας αυτονομία. Το αντίθετο συμβαίνει. Έχουμε πολλές τον έλεγχο της ασφάλειας του εφοδιασμού συχνά διότι υπάρχει ε, αυτό το πολιτικό σκέλος ε, και με τις ε, ιδιωτικοποίησεις, αποκρατικοποίησεις χάνουμε τον έλεγχο του εφοδιασμού στην Ευρώπη. Επίσης χάνουμε τον έλεγχο στρατηγικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών στρατηγικού χαρακτήρα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ε, Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, για τον εξοπλισμό και προφανέστατα χρειαζόμαστε και τη διαφάνεια. Πώς να λειτουργήσει εύρυθμα η αγορά ε, εάν συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο γίνεται κατασπατάληση των πόρων από τις κυβερνήσεις, ενώ λόγω των εξελίξεων χρειαζόμαστε αυξανόμενη διαφάνεια ακριβώς για να μεριμνήσουμε ώστε ε, να είναι ε, πιο χρηστή η διαχείριση των πόρων και όχι μόνο αυτό, αλλά και συγκέντρωση και κοινή χρήση των πόρων μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε στρατηγικό σχεδιασμό, διαλειτουργικότητα πάλι για να αξιοποιήσουμε καλύτερα ε, την εισφορά των φορολογουμένων και να καλύψουμε τις ανάγκες μας ε, ως προς την ασφάλεια και την άμυνα. Νομίζω πως ε, τα αφήνουμε σε μεγάλο βαθμό όλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ρόλο και αυτός είναι ένας από τους στόχους της έκθεσης, πέραν από το να τροφοδοτήσουμε την αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την υλοποίηση των οδηγιών του πακέτου, του αμυντικού πακέτου, με, επί τη βάση στοιχείων που θα προσκομίσουν τα κράτη-μέλη. Δεν αμφιβάλλω για αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δούμε την έκθεση, αλλά πρόσφατα, επειδή ξέρω πολύ καλά μια συγκεκριμένη περίπτωση στη χώρα μου, την, ε, έκανα μια ερώτηση για την επαναδιαπραγμάτευση των αντισταθμιστικών οφειλών για αγορές, ε, στρατιωτικές προμήθειε για τις αντισταθμιστικές ε, οφειλές ε, που υπήρχαν ε, Ήδη όταν τέθησαν σε ισχύ αυτές οι οδηγίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε καν παρατήρησε ότι είναι, ε, σημειώνεται μια κατάφορη ε, παραβίαση αυτών των ε, διγιών με τα υποβρύχια και την επαναδιαπραγμάτευση των αντισταθμιστικών οφειλών και έγραψε στην αρμόδια επίτροπο, έκανε και στον προκάτοχό του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως η οποία υποτίθεται ότι λειτουργεί ως θεματοφύλακας και φροντίζει να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη σωστά αυτές τις οδηγίες, ε, δεν ε, αντιδρά. Θα καταθέσω τροπολογία στη δική μου την έκθεση, διότι γνωρίζετε τους περιορισμούς που υπάρχουν ως προς τον αριθμό των λέξεων. Και ο εισηγητής ε, κάνει ένα πρώτο σχέδιο και στη συνέχεια τροποποιεί με τροπολογίες κάποια σημεία ή διευρύνει, το, ε, ε, επεκτείνει το πεδίο. Επίσης θα καταθέσω τροπολογίες για το σχέδιο της Σύμκο, που εστιάζεται περισσότερο ε, στο νομοθετικό κομμάτι και ελπίζω να υιοθετηθούν οι τροπολογίες μας από, τις, από τους συναδέλφους ε, της ΙΜΚΟ. <clears throat> Δεν είμαι σίγουρη αν είναι εδώ ο συνάδελφος από την ΙΜΚΟ. Νομίζω ότι είναι συμπληρωματικό το σχέδιο της ΙΜΚΟ σε σχέση με ε, τα στοιχεία που ε, πραγματεύομαι εγώ μέσα στην έκθεσή μου και έτσι θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να εισακουστεί η άποψη του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο του Ιουνίου για το ίδιο ζήτημα. Τέλος, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδρου Κερέιρα που θα κάνει την έρευνα ε, και θα στάξει την έκθεση και τον Μισελ Γιαρασέκ από την Γραμματεία που βοήθησε ουσιαστικότατα με τη συμβολή του σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε. Η συγγήτρια της ΕΜΚΟ είναι η κυρία Κάπετς, η οποία θα βρίσκεται εδώ σε λίγα λεπτά, ελπίζουμε, και θα ακούσουμε και τα όσα έχει να μας πει η ίδια. Να δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Όπως καταλαβαίνω, απουσία του κύριου Κίρτσου, ο κύριος Γκάλαρ θα πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, πράγματι ο κύριος Κίρτσος δεν κατάφερε να βρίσκεται εδώ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας ε, και την πολλή δουλειά που κάνατε. Το σχέδιο αυτό είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση περιγράφοντας την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά. Αναφέρατε την έλλειψη συντονισμού, την έλλειψη ε, ε ομοιομορφίας ε, που υπονομεύει τη στρατηγική μας αυτονομία και αποδεινώνεται λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι αμυντικές μας αγορές είναι σημαντικές. Ε, παρέχουν ε, θέσεις εργασίας εξειδικευμένες ε, στην Ευρώπη και είναι σημαντικές και για άλλους τομείς της οικονομίας όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, οι τεχνολογίες διπλής χρήσης και οι συνέργειες μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών τεχνολογιών επηρεάζουν επίσης σε κάποιο βαθμό την ανάπτυξη. επειδή πρόκειται φυσικά για ένα στρατηγικό τομέα, δεν ε, λειτουργεί με ε, βάση μόνο του κέρδους. Διότι αν συνέβαινε αυτό δεν χρειαζόταν να σκεφτόμαστε τους περιορισμούς εξαγωγών όπλων, ούτε να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί, ούτε να θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατές αγορές ε. αλλά οι πολιτικές συνθήκες μας επιβάλλουν άλλα. Ο ισχυρός συζητητής ε, λέει ότι θα προτιμούσε μια πιο ακριβή επισκόψη της καταστάσης εφαρμογής ε, των ε, πακέτων για την άμυνα. Υπάρχουν σχετικές παράγραφοι. Εμείς θέλουμε μια πιο ολοκληρωμένη επισκόψη του τμήματος της έκθεσης όπου συζητείται σαφώς ποιες ήταν οι προθέσεις, τι ακριβώς έχει επιτευχθεί και τι όχι. και φυσικά θα μας βοηθήσει να γνωρίζουμε τι έχει επιτευχθεί. Όπως και σε άλλους τομείς. Ειδικότερα εδώ ε, κρίσιμη σημασία έχει η πολιτική βούληση των κρατών μελών ώστε να σημειωθεί κάποιο πρόοδος. Επίσης ε, αναφέρεται και στη δική μου έκθεση ως και ε, στην έκθεσή μου του Οκτωβρίου 2013 για την Ευρωπαϊκή ε, Βιομηχανική Βάση Τεχνολογίας και Άμυνας και συγκρίνει τα όσα υπόθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής Δεκεμβρίου του 2013 και τη σημερινή κατάσταση. Πόσο έχει εφαρμοστεί πλήρως και σωστά η υλοποίηση αυτών των δύο ε, οδηγιών. θα αποτελέσει πολύ καλή συμβολή πιστεύω η έκθεση αυτή για τη Σύνοδο Κορυφής ε, για την άμυνα. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα σχόλια για την παράγραφο 4 όπου αναφέρεται σε αυξημένη ε, επένδυση. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, ε, ίσως να μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, αλλά έτσι όπως αναφέρετε, να πω, υπάρχει όντως αυξημένη ξένη επένδυση στο τομέα της άμυνας. Στην παράγραφο 9 αναρωτιόμαστε κατά πόσο χρειαζόμαστε γενικά κίνητρα για να αυξηθεί η ελκυστικότητα των έργων συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο ακριβείς να ζητήσουμε κίνητρα για διεθνή συνεργασία εντός της ΕΝΤΑ και της ΟΚΑΡ σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες των φοροαπολαγών για οργανισμούς ε, υποστηρικτικούς του ΝΑΤΟ. Αλλά το να λέμε απλά φορολογικά κίνητρα για αυξημένη συνεργασία Φυσικά όλοι κινούνται περισσότερο όταν υπάρχουν επιπλέον φορολογικά κίνητρα. Αρκεί να μην ε, κοστίζει υπερβολικά πολύ η εφαρμογή του και να χρειάζονται επιπλέον κρατικά κονδύλια. Για την παράγραφο 11. αναρωτιόμαστε κατά πόσο υπάρχει όντως αυξημένος κίνδυνος παραβίασης της κοινής θέσης ε, ε, για τις εξαγωγές όπλων. Είναι τόσο εμφανέ ότι τέτοιε άδειε εξαγωγή όπλων χρησιμοποιούνται από κράτη-μέλη ω ε, εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε ένα ερωτηματικό. Και εδώ Ολοκληρώνεται τα σχολεία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλα. Να δω τώρα κατά πόσο θα έχουμε τη συμμετοχή των σκιωδών ή των εκπροσώπων τους και από όσο κατάλαβα η κυρία Λέζινγκ να σκιώδη συγγήτρια. Οπότε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όλα βασίζονται σε μια πεποίθηση που θεωρείται προφανής για όλες τις περαιτέρω προτάσεις και αναλύσεις. Αλλά εγώ την αμφισβητώ. Πάντα θεωρούμε όσο λιγότερα χρήματα υπάρχουν για την άμυνα στην ε, Ένωση και στους εθνικούς προπολογισμού, ότι μάλλον είναι αυταπόδεικτο ότι ο, παντού έχουν γίνει περικοπές στους αμυντικούς προπολογισμού. Ναι, αυτό μπορεί να ισχύει σε κάποιες χώρες. Βεβαίως, σε ορισμένες χώρες έχουν μειωθεί λιγάκι, αλλά μεταξύ 2000 και 2013 από 270 δις σύμφωνα με την ανάλυση του Τσίπρη, στα 279 δις. Άρα δεν ισχύει η βασική μας προϋπόθεση ότι μειώνονται οι αμυντικές δαπάνες. Και γι' αυτό όμως απαιτούνται όλο και περισσότερα. Θέλουμε να βελτιωθούν οι δυνατότητές μας ε, στρατιωτικής παρέμβασης. Λέμε πάντοτε θέλουμε να υπάρχει περισσότερη συνεργασία για να εξοικονομήσουμε χρήματα των φορολογουμένων όπως ε, συχνά λένε τα μέσα. Βεβαίως, ε, αν αυτά πρόκειται κατόπιν να δαπανηθούν στο κοινωνικό τομέα συμφωνώ, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η πρόθεση. Και να με πείσετε ότι δεν ισχύει αυτό αν μπορείτε. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που για μένα είναι ιδιαίτερως προβληματικά. Και για άλλους τομείς λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια σχεδιασμού. Διότι και εδώ τίθεται θέμα ότι δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να ελέγχουν ε, την κατάσταση. Ορισμένοι λένε μάλιστα ότι οι έλεγχοι από τα κράτη-μέλη δημιουργούν πρόβλημα. Πουθενά δεν έχω ακούσει ότι πρέπει να βελτιωθεί αντίστροφα η δυνατότητα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα, καλύτερο σχεδιασμό σημαίνει λιγότερη δημοκρατία. Αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνη. Να δώσουμε και άλλες φοροαπαλλαγές για συνεργασίες στον τομέα της ε, άμυνας και των εξοπλισμών. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό φοροελαφρύνσεις για τη βιομηχανία εξοπλισμών είναι στην ουσία επιδοτήσεις για τις βιομηχανίες όπλων. Και αυτό το απορρίπτουμε. Επίσης, η έκθεση αυτή θέλει να δημιουργήσει έναν στρατιωτικό βιομηχανικό κλάδο. Αλλά η πείρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες καταδεικνύουν ότι η δημιουργία ενός τέτοιου τομέα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να το επανεξετάσουμε, να μάθουμε από την πύρα Για τις εξαγωγές όπλων το ανέφερε και ο κύριος Γκάλερτ. Συμφωνώ και συμμερίζομαι με τις ανησυχίες του, γιατί σε τελευταία ανάλυση οι εξαγωγές όπλων είναι πάντα πολύ επικερδείς για τον κλάδο αυτό και συμμερίζομαι τις ανησυχίες του ότι βραχυπρόθεσμα δεν θα βελτιωθεί ο έλεγχος ακριβώς των εξαγωγών. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για τους οποίους απορρίπτει η ομάδα μου την έκθεση αυτή και για το θέμα αυτό θα υποβάλουμε έκθεση μειοψηφίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Έφτασε μόλις ο κύριος Μπιτικόφερ, ε, σκιώδης για τους πράσινους. Ε, θέλετε το λόγο. Εάν μου τον δίνετε, Πρόεδρε, πολύ ευχαρίστως. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και κάποιες ειδικότερε. Η πρώτη γενική παρατήρησή μου είναι πως ήμουν ανέκαθεν κατά της αρχής που προβάλλεται μέσα σε αυτή την έκθεση το τέστην ότι ε, η, Ευρωπαϊκή Ένωση τάσεται υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας. Αυτή, αυτό το δόγμα στο Β ή στην πρώτη παράγραφο είναι γελίο. Είναι αδιανόητο να προκύψει κάτι που με ειλικρίνεια θα εξασφαλίζει συμμόρφωση με τα κριτήρια. Αν πραγματικά ειλικρινά Θέλετε να μιλήσετε για στρατηγική αυτονομία. Ίσως στο παρελθόν να ήταν δυνατό αυτό, όμως στη σήμερον ημέρα και για να είμαστε ρεαλιστές δεν μπορούμε να επιδιώκουμε ιδεολειψίες, ε, ιδεολογικού χαρακτήρα στόχους. Ε, δεν πρόκειται η ευρωπαϊκή ασφάλεια να κατοχυρωθεί αποκλειστικά και μόνο από θεσμικά όργανα της Ένωσης μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να ε, στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας να ενισχύσει το ρόλο της, δεν είμαι κατά αυτού. Όμως είναι ε, ουτοπική η ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας και θα πρέπει να σταματήσουμε να κυνηγούμε αυτή τη χήμερα. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι αντιφατικό πως μέσα στην έκθεση αυτή αφενός εκφράζουμε τη λύπη μας ε, για τις υπερβολικές δαπάνες στην Ευρώπη και να πω εδώ ότι Είμαστε στη δεύτερη θέση παγκοσμίω όλοι μαζί, τα 28 ε, κράτη-μέλη της Ένωσης, με 190 δις. Σε... Είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει λοιπόν να μειωθεί αυτό το ποσό και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων και μέσα στην έκθεση επαναλαμβάνουμε το ότι θα δώσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και μάλιστα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με συστηματικό τρόπο ε, ε, τα σώταν κατά αυτού η ομάδα μου στο παρελθόν και εξακολουθούμε να το πιστεύουμε το μόνο που θα συμβεί είναι να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία να αντλεί χρήματα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αντί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και αυτό είναι ένα πρόσχημα για να μην επιτευχθεί στον, ε, σε ικανοποιητικό βαθμό το pooling and sharing, αυτή η ομαδοποίηση και ε, κοινή χρήση των πόρων. Τρίτον, δεν πιστεύω πως ε, είναι σωστό να δίνουμε φορολογικά κίνητρα και μιλώ για την παράγραφο 9 εδώ Φορολογικά κίνητρα λοιπόν για το pooling και sharing. Ε, μιλούμε για ευημερία της ε, βιομηχανίας. Όχι, ο στόχος είναι να είμαστε λογικοί και να επιτύχουμε μια χρήστη χρήση των κονδυλίων, pooling and sharing. Βεβαίως, για πολιτικούς λόγους είμαστε 200% υπέρ, όχι όμως με κατάχρηση των πόρων που προέρχονται από τους ε, φόρους. και δεν μπορούμε να ε, ε, υποστηρίξουμε μια έκθεση που έχει μια τέτοια διάταξη. Τέταρτον, στο παρελθόν έχω διαφωνήσει με την εισηγήτρια όταν κατέθεσε μια έκθεση για την θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε την είχα επικρίνει και το επαναλαμβάνω εδώ διότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί ότι μπορεί να έχει το ρόλο του παγκοσμίου παρόχου ε, ασφάλειας. Εδώ δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα δικά μας ή να, να, να, ε, ε, εξάγουμε την ασφάλεια, αν θέλετε, στις άμεσα γειτονικέ μας χώρες. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αναλάβουμε τέτοιο ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αυτή την έκθεση βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται στρατηγικές ως όμοιροι. Δηλαδή, αναφέρομαι στην ε, στρατηγική του pooling and sharing, που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Και, ε, περιπτώσει, ας αποφασίσουμε αν θα συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας, αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη ή εάν ε, υποστηρίζουμε αποκλίνουσες πολιτικές οι οποίες συνεπάγονται ότι ε, πάνω στην κοινή πλατφόρμα θα προσπαθήσουμε να χώσουμε και άλλα πράγματα που εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα, όπως παίρνοντα το παράδειγμα ε, της ομοιρίας του pooling and sharing, στο οποίο προαναφέρθηκα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί η πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είμαστε αρνητικοί. Θα χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που έχουμε να ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση, διότι με τα χαράς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αν ο στόχος είναι να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο, οφείλω να ομολογήσω, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μία ιδεολογική ρότα που ε, έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν κάποιοι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Από σου καταλαβαίνω δεν υπάρχουν... Α, ζήτησε το λόγο ο κύριος Γκάλερ. Ναι, να απαντήσω σε ορισμένα σημεία. Για τα αριθμητικά στοιχεία, αγαπητοί συνάδελφοι Λέζινγκ, τα στοιχεία του Τσίπρη, αν δούμε αυτά τα 270 και 279 δις, δεν ξέρω ούτως ή άλλως με ποια ισοτιμία έχει υπολογιστεί αυτό μεταξύ του 2000 και του 2013. Ποιο ήταν το δεύτερο στοιχείο, 2000 και 2013. Ε, κυρία Λόιζινγκ, μιλάει χωρίς μικρόφωνο. 2000 και 2013, δεν είπατε συνεχίζει ο κύριος Γκάλα. Ναι. Θα ήταν ε, ούτως ή άλλως ενδιαφέρον να δούμε με τι ισοτιμία και σε ποιο νόμισμα και να δούμε και τον πληθωρισμό. Και με τον ε, πληθωρισμό ίσως να είναι και μείωση. Ε, με τα δικά μου στοιχεία τουλάχιστον σαφώς υπάρχει μείωση των αμυντικών προϋπολογισμών. Και πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αλλαγή στην κατάσταση πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Την, την αλλαγή στην κατάσταση ασφάλειας και άμυνας. Και πρέπει να δούμε εάν επιτέλους θα δημιουργήσουμε το δικό μας ανεξάρτητο δυναμικό να μπορούμε να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις ή θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξαρτώμεθα από τον Α στη μία περίπτωση, από το Β στην άλλη περίπτωση. Οπότε δεν είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε μαζί από κοινού και να έχουμε αξιόπιστη αποτροπή, δυνατότητα αποτροπής μόνοι μας. Το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας. Όταν ακριβώς ε, βρίσκεται για, ε, πρόκειται για γειτονικές μας περιοχές, θεωρώ ότι έχει και την εξής άποψη. Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα πούμε εντάξει, πρέπει να αναλάβουμε κάτι με μια γειτονική μας χώρα και μετά πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα το ΝΑΤΟ και μετά η Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ να πει όχι χρειάζεται ομοφωνία, εγώ δεν συμφωνώ για το τάδε για τη Συρία την Τουρκία ή την Λιβύη. Θα πρέπει να έχουμε αυτόνομη δυνατότητα δράσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό και για την ε, γειτονική μας περιοχή είναι σημαντικό να μπορούμε να το πράξουμε. ούτω ώστε να μην μπορούν κάποιοι εκτό τη Ένωση να έχουν δικαίωμα βέτο στη δράση μα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντρογεύσκη. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι έχει εξαιρετική δομή και διατύπωση η έκθεση, δεν είναι πολύ μεγάλη, επισημαίνει τα σημαντικότερα ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα δύο σχόλια για κάποια πράγματα που θεωρώ ότι λείπουν αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, πρέπει πιστεύω να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την έκθεση. Γνωρίζουμε φυσικά ότι οι δαπάνες και η εξέλιξή τους ε, δημιουργούν ανησυχίε. Στο πρώτο μέρος της έκθεση για την ανάπτυξη των ε, αμυντικών αγορών και για τους κινδύνους ε, της αυτονομίας. Το σημείο 1 γίνεται παραγραφό 3 και υπάρχουν και άλλε αλλαγέ ε, και με αυτή τη λογική θα αναφέρομαι σε μεγαλύτερε απειλέ και να είναι πιο λογική η σειρά. Το δεύτερο αφορά τις αντισταθμιστικέ οφειλές. Ε, εγώ υπήρξα μέλος της ε, σχετικής επιτροπής και κάθε χρόνο είμαστε όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά το πρόγραμμα αντισταθμιστικών οφειλών, όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και για τις άλλες χώρες. Μου κάνει έκπληξη λοιπόν που εξακολουθούμε να συμπεριλαμβάνουμε αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουμε ήδη πιστεί ότι τα θέλουμε. Και μετά ε, ε, μια παράκληση. Είμαι επιφυλακτικός όσον αφορά ορισμένα στατιστικά στοιχεία. Παλιότερα ήταν εύκολο να αξιολογήσει κανείς ε, τις αμυντικές δαπάνες. Αν αυτές αυξάνονταν, είχαμε καλύτερη άμυνα, αλλά πολύ συχνά στον αμυντικό τομέα, στην αμυντική βιομηχανία. Ε, μου λένε διάφοροι εμπειρογνώμονες ε, ε, ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες στο στρατιωτικό τομέα, στον αμυντικό τομέα και μου δείχνουν τον προπολογισμό τους και όταν βλέπω τα νούμερα εκεί ανησυχώ ακόμη περισσότερο. Οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται και απόψη ποιότητα. Δεν είναι μόνο θέμα ποσοτήτων. Ε, δεν είναι μόνο οι ποσότητες που βλέπετε στον προπολογισμό. Πρέπει να δούμε και κατά πόσο οι δαπανε παρέχουν πράγματι καλύτερη ασφάλεια και κατά πόσο αυτά τα ουσιώδη στοιχεία βελτιώνουν ή την κατάσταση. Έχουμε του προπολογισμού μα όπου πρέπει να δαπανούμε περισσότερα σε στρατιωτικέ συντάξει. Για παράδειγμα, αυτέ οι δαπάνε αυξάνονται. Ε, χωρίς να βελτιώνεται κάτι. Ενώ πρέπει να, ας πούμε, αναπτύξουμε την τηλεματική. Σε ορισμένους τομείς ε, δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να έχουμε τις ε, νεότερες τεχνολογίες που θα βελτίωναν την απόκρισή μας σε ορισμένες καταστάσεις. Και συμφωνώ και με τον κύριο Αγκάλαρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόφερ, Ζητήσατε το λόγο για τη δεύτερη φορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στα όσα είπε ο κύριος Γκάλαρ. Κύριε Γκάλαρ, αντιλαμβάνομαι την επιχειρηματολογία σας, την πιστεύω, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή αιτιολογεί τη διατύπωση στρατηγική αυτονομία. Αυτό που θα δεχόμουν θα ήταν κάποια διατύπωση που να λέει ενισχυμένες στρατηγικές ευθύνες ή ενισχυμένες ε, στρατηγικές ε, δυνατότητες, διότι ναι, έχουμε μεγαλύτερο βάρος να αντιμετωπίσουμε, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ή να δημιουργήσουμε ε, την εντύπωση ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε όλο το βάρος εμείς. Για ορισμένα ζητήματα, ναι, η Ευρώπη θα μπορούσε να δράσει μόνη, ίσως, ίσως έχει δράσει μόνη της, ίσως όχι επιτυχώς ή ίσως όχι με επαρκή επιτυχία, αλλά η στρατηγική αυτονομία είναι μια πολύ ευρεία έννοια που όπως την καταλαβαίνω εγώ εννοεί ότι θεωρητικά θα έπρεπε να μπορούμε να δράμε μόνοι μας κάθε φορά που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο ή αποφελές οτιδήποτε. Και κατά με κάτι τέτοιο που θεωρουμε οτι ειναι απαραιτητο η αποφελες οτιδηποτε και κατα κατι τετοιο ειναι μη ρεαλιστικό και περιλαμβάνει και τις σχέσεις ασφαλείας μεταξύ παράδειγμα της Ευρώπης και, ε, και των ΗΠΑ. Ουσιαστικά παραβλέπει ε, εταιρικές σχέσεις στον τομέα της ασφαλείας που έχουμε με άλλους εταίρους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτό το διέξοδο. Για να διατυπώσουμε αυτό που λέτε, μπορούμε να βρούμε μια διατύπωση την οποία θα στηρίξω και εγώ. Η άλλη παρατηρήση που θέλω να κάνω, να επαναλάβω, όταν μιλάμε για 190 δις τα οποία δαπανώνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εποχές όπου όλοι γυρνούν στην παλιά συνήθεια του να ζητούν επίπεδο του 2% του ΑΕΠ ε, για τις χώρες μας. Εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να ε, τονίσουμε την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και των δαπανών. Και όχι ε, ένα απλό ποσό. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια της Ευρώπης, επιμένοντας για περισσότερη ποιότητα και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Και αυτό φυσικά σημαίνει το να ομαδοποιήσουμε ε, και τις δυνάμεις της αγοράς ε, χωρίς να αφήνουμε τον καθένα στο δικό του τμήμα, στη δική του πλευρά σε μια αγορά κατακαιρματισμένη ε, στο παρελθόν έχει σημειωθεί πρόοδος υποστηριζόμενη από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου εδώ για να, για να διευρυνθεί η αμυντική αγορά. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο μεγάλη τελικά αυτή η αγορά. Αν την μεταμορφώσουμε όμως σε μια λειτουργική αγορά, τόσο πιο περισσότερο ε, εποφελής θα είναι για τους πολίτες ε, και τόσο περισσότερο θα ενισχύσει την ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτό πιστεύω πρέπει να τονίσουμε. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκόμες, για άλλη μια φορά έχετε το λόγο για να σχολιάσετε ή να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ίσως ε, Αφού απαντήσω, θα ήθελε και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ή η Επιτροπή να σχολιάσουν, ε, διότι τους ενδιαφέρουν πολλά από τα σημεία που αναφέρθηκαν στη ζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, μου πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γκάλλαρ. Αναφέρομαι στις ξένες επενδύσεις, ε, διότι αυτό μου λένε ότι συμβαίνει. Ίσως όχι σε όλες τις χώρες, αλλά σίγουρα σε κάποιες, ε, κυρίως αυτές που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, όχι μόνο για εκείνες τις χώρες, αλλά και για το μέλλον της ε, ευρωπαϊκής άμυνας, διότι ορισμένες φορές μιλάμε για επενδύσεις που σχετίζονται με τεχνολογικές εξελίξεις σε λίγα στρατηγικούς τομείς, όπως παραδείγματος χάρη διάστημα, ε, ασφάλεια, θαλάσσια ασφάλεια και αυτό δεν συμβαίνει μόνο για τα κέρδη δεν είναι μόνο γι' αυτό που κάποιοι ξένοι επενδυτές εξαγοράζουν ε, τέτοιες ε, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Συμβαίνει αυτό, ίσως όχι σε όλες τις χώρες, ξαναλέω. Πάντως θα ήταν θλιβερό να παραγνωρίσουμε τη σημασία αυτής της εξέλιξης και ξαναλέω, θα πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό όταν εξετάζουμε το θέμα γενικότερα. Για τις αντισταθμιστικές οφειλές ε, ένα άλλο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Γκάλερ και άλλοι συνάδελφοι είναι αυτό των φορολογικών κινήτρων για τις πρωτοβουλίες pooling and sharing. Ε, εγώ υποστηρίζω αυτή την ιδέα, ίσως κάποιοι διαφωνούν και σέβομαι τους λόγους για τους οποίους διαφωνούν, όμως εγώ εξακολουθώ να την υποστηρίζω την ιδέα, διότι έχουμε, ε, ε, συζητάμε εδώ και τόσο καιρό αυτή την πρωτοβουλία, αλλά δεν σημαίνει ποτέ τίποτα. Το Βέλγιο, από ό,τι μου είπανε, πρόσφατα αποφάσισε σε, στα πλαίσια μιας τέτοιας πρωτοβουλίας ε, να χρησιμοποιήσει αυτή την εξαίρεση και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στον τομέα αυτό διότι δεν έχουμε υπάρξει ε, αποτελεσματική σε σχέση με το ε, να περάσουμε στην πράξη μετά από τα λόγια είτε μιλάμε για χώρες που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ είτε όχι. Είναι κέρυες σημασία στο ζήτημα διότι είναι πενιχροί οι πόροι ή φορολογούμενοι δικαίως περιμένουν καλύτερα κριτήρια ε, για, την, ε, για τις αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των πόρων στον τομέα της άμυνας Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν περιττές δαπάνες λοιπόν, καμία επικάλυψη. Αυτό μόνο μέσω της ομαδοποίησης και κοινή χρήση των πόρων μπορεί να συμβεί με την κοινή έρευνα, την ε, κοινή χρήση τεχνολογιών εχμής και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο στόχος των φορολογικών κινήτρων. Θα υπάρχουν και άλλα κίνητρα, είναι ένα μόνο παράδειγμα, αλλά είναι σημαντικό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, θα εποπτεύει τη διαδικασία και παρεπιπτόντος να σας πω πως θα πρέπει να βασιστούμε στα στοιχεία ε, που συλλέγεται ώστε να μην ε, είναι μόνο βραχυπρόθεσμη προσέγγιση μας αλλά και μακροπρόθεσμα αξιολογούμε τις στρατηγικές μας ανάγκες. Τώρα, ο κύριος Γκάλερ και συμφωνώ μαζί του και γι' αυτό το αναφέρω μας είπε πως η κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων, μάλλον δεν ξέρω και αν συμφωνώ απολύτως μαζί του ή αν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε. Νομίζω όμως πως σε σχέση με αυτά που έχω ήδη γράψει στην έκθεση θα μπορέσω σε συνεργασία με τους σκιώδους συζητητές να επεκταθώ διότι σε αυτό το τομέα βλέπουμε ότι δεν έχουν δείξει ιδιαίτερη σοβαρότητα ε, τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, ε, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ για την Λιβύη παρουσίασε μια έκθεση, μιλούσαμε για τις εξαγωγές όπλων και δύο κράτη-μέλη μαζί με άλλα κράτη ήταν στον κατάλογο αυτών που πουλούσαν όπλα παρά το εμπάργο, την απαγόρευση εξαγωγών, παρά ε, το ότι ε, υπάρχει πληθώρα προβλημάτων όπως η τρομοκρατία στη χώρα, εσωτερικές συγκρούσεις κτλ. Οπότε σίγουρα δεν ε, κάνουν καλά τη δουλειά τους τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικότατο ρόλο για την υιοθέτηση αυτής της κοινή θέση, οπότε θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση της εφαρμογής από πλευράς των κρατών μελών και αυτό θα έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος όταν, μιλούμε, όταν αρχίσει η συζήτηση για την αξιολόγηση εφαρμογής των οδηγιών του αμυντικού πακέτου. Ε, κυρία Λέζιν, ίσως μπορούμε μπορούμε, ίσως ε, μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με το πού διοχετεύονται τα κονδύλια και θα δω τα συγκεκριμένα στοιχεία διότι ενδέχεται σε ορισμένε ε, περιπτώσεις να είναι υπερβολικές ε, οι δαπάνες να... ή να υπάρχουν δαπάνες που δεν ενισχύουν το αμυντικό δυναμικό. Παραδείγματος χάρη, δύο κράτη-μέλη έχουν υπερβολικές δαπάνες για την, ε, τα πυρηνικά τους όπλα. Ε, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν ενισχύει, το αντίθετο μάλιστα, την, ε, το αμυντικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα πρέπει να το δούμε και κατά αναλογία σε σχέση με το συνολικό ποσό των αμυντικών δαπανών. Αντίθετα υπάρχουν ε, λιγοστές δαπάνες σε τομείς που χρειαζόμαστε περισσότερο δυναμικό. Το χρειαζόμαστε ούτω ώστε οι στρατιώτες μας, οι γυναίκες και οι άντρες ε, μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, ε, να διαφυλάξουν τη ζωή τους και να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πώς δαπανούμε τα κονδύλια, ποιες δαπάνες είναι καλές, ποιες είναι κακές σε σχέση με τις αμυντικές μας ανάγκες, διότι ναι, στόχος είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε τα κονδύλια. Προτού τα αυξήσουμε και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το αμυντικό πακέτο, διότι συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν πολύ μεγάλη διαφθορά. Η αδιαφάνεια, το ύψος των κακών δαπανών, η στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, διότι δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις ενίας αγοράς. Κύριε Μπιτικόφερ, νομίζω αναφέρθηκα ήδη σε κάποια από τα ζητήματα που θέσατε. Εξακολουθώ να σέβομαι την απόψή σας, δεν συμφωνώ όμως καθόλου με αυτό που είπατε ότι είναι γελία η αρχή της στρατηγικής αυτονομίας, δεν την εφήβρα εξολογώ, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης και άρα πιστεύω ότι χρειαζόμαστε στρατηγική αυτονομία για κάποια βασικά ζητήματα. Παραδείγματο χάρη, δεν θέλω να έχω να περιμένω τους Αμερικανούς να πατήσουν το, το κουμπί για να αποφασίσουν αν εγώ θα έχω GPS ή όχι ή ε, να περιμένω από μια κινέζικη επιχείρηση που ε, ελέγχει τι βασικές τεχνολογίες για την κυβερνοασφάλειά μας. Εγώ δεν θέλω να εξαρτώμαι από αυτούς. Αν αυτό θέλει ο κύριος Μπιουτικόφρη, πρόβλημά του. Εγώ πάντως ε, πιστεύω ότι πρέπει εμείς να φροντίσουμε τα περιστρατηγικής αυτονομίας μας στον τομέα της αμυντικής ε, βιομηχανίας όπου πραγματικά το χρειαζόμαστε και γι' αυτό ακριβώς ε, αυτό θα πρέπει να τονίσουμε και να περάσει αυτό στην ανάλυση που θα γίνει για την εφαρμογή του πακέτου, του, του αμυντικού πακέτου. Δεν πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια θα είναι φυσικά θέμα και θα το αναλάβουν μόνο οι θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν γέλιο και ε, δεν το περιμένουμε. Υπάρχουν δύο κράτη-μέλη που θα ε, εξακολουθήσουν να έχουν το σημαντικότατο ρόλο που έχουν σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η συνεργασία. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν κάνουν καν το ελάχιστο. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το ελάχιστο δεν κάνουν σε σχέση με τις ε, κείμενες συνθήκες ε, όταν πήγαμε στο Βόρειο Ιράκ είδα ότι τα κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνταν στο, στο στρατιωτικό τομέα υποστήριξη των Πασμέργα ε, των Κούρδων δεν ε, συντονίζανε τη δράση τους. Ε, Είχαν εξοπλισμό. Είχαμε εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τους Πεσμέργα εάν υπήρχε καλύτερος συντονισμός. Ε, θα συμφωνήσετε, δεν μπορεί κύριε Μπιουτικόφερ, ότι ε, είναι σημαντικό αυτό ε, στο βασικότερο μέτωπο που έχουμε παραδείγματο χάρη η καταπολέμηση του ISIS στο Ιράκ. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους στα κράτη-μέλη, διότι ακριβώς δεν ενώνουν τις δυνάμεις τους, δεν συνδυάζουν τις προσπάθειες προσπάθειές τους δεν συντονίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό έχουμε την είπατε εκπρόσωπο για την ε, ε, κοινή εξωτερική πολιτική και η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας είναι μέρος εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων γιατί μιλάτε ε, κύριε Μπιουτικόφερ για την ε, ορθολογική χρήση ε, των χρημάτων των φορολογουμένων και φυσικά συμμερίζομαι την ανησυχία σας. Για πείτε μου λοιπόν τι κάνετε στην ε, με τη διαφθορά ε, που ε, που στη διαφθορά στις συναλλαγές ανάμεσα στα κράτη-μέλη η χώρα σας και η χώρα μου παραδείγματος χάρη και γι' αυτό σας λέω ότι είναι σημαντικό να γίνει ανάλυση της εφαρμογής του πακέτου των αμυντικών οδηγιών γιατί αυτό θα επιφέρει ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας για να πάψει επιτέλους αυτή η διαφθορά και έτσι Ε, θα βγω αληθινής σε αυτά ε, που έχω πολλά σε επί δημοσίως, αλλά δεν με έχουν υποστηρίξει οι συνάδελφοι. Τέλος, τέλος. Για τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Το θέμα που ο συνάδελφος ε, Ζωροβιεύσκη. Ναι, οπωσδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Εδώ είδαμε ότι υπάρχει διαφορετική άποψη μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας όταν πέρναγε το πακέτο για την άμυνα. Η Επιτροπή υποτίθεται ότι είναι κατά των αντισταθμιστικών ε, ωφελών. Αλλά στην ουσία δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Ο ίδιος ο Επίτροπος ε, Φεστχάγκερ είχε πει ότι δεν τον ενδιαφέρε. Όταν συζητάγαμε μια ανεδιαπραγμάτευση ενός συμβουλαίου, συμβολέου του 4 το 14. Σαφώς δηλαδή μετά την ε, θέση σε ισχύ του, του πακέτου άμυνας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Άμυνας είχε και νομίζω ακόμη έχει διαφορετική προσέγγιση. Αναγνωρίζει τη σημασία των αντισταθμιστικών ωφελών εφόσον τα ωφέλη αυτά στοχεύουν να, ε, να ενισχύσουν την αμυντική δυνατότητα και να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή τεχνολογική και αμυντική βάση. Να δούμε αν έχουν ε, μειωθεί διαφορές αυτών των απόψεων. Θα υποβάλω τροπολογίες για αυτό το θέμα στην έκθεση της ΙΜΚΟ. γιατί δεν μπορώ να υποβάλω όσα κειμένα θέλω, υπάρχουν περιορισμοί. Αλλά θα μπορούσε να ενταχθεί στην έκθεση ΙΜΚΟ, γιατί αφορά περισσότερο τις νομοθετικές πλευρές. Αλλά καλωσορίζω τροπολογίες και από τους συναδέλφους γι' αυτό και είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ με όλους που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια να καταλήξουμε σε μία αποδεκτή κατάληξη για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την αποτίμηση της Κομισιόν και τις συζητήσεις του Συμβουλίου και ελπίζω να καταλήξουμε και σε δράση. Ευχαριστούμε. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών τόσο στην ΣΕΝΤΕ όσο και στην ΕΜΚΟ είναι η τελευταία ημέρα του Μαρτίου. 31η Μαρτίου στις 12 η ώρα. Σε συνιστώ να τηρήσετε τη όρια των αρμοδιοτήτων των δύο επιτροπών κατά την υποβολή τροπολογιών. Επόμενη εξέταση στις 6 Μαΐου. Ε, εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο και περνάμε στα διάφορα. Υπάρχουν αιτήματα. Όχι. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, απογευματινή συνάντηση, όπου θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ιαν Στόλτεμπεργκ, και στη συνέχεια θα βρίσκεται ο συντονιστής αντιμετώπισης τρομοκρατίας, ο κ. Κακόφ. Κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ και ΣΕΝΤΕ. Επόμενη συνεδρίαση της ΣΕΝΤΕ έχει προβλεφθεί για τις 16 Απριλίου. Ευχαριστούμε πολύ για την διήμερη συνάντηση. Να ζητήσω από τους συντονιστές και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να παραμείνουν για το διευρυμένο Προεδρείο.